Äh, Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση στην έναρξη της συνεδρίασης από όλους τους παρευρισκόμενους και από όλους τους διερμηνείς που ήρθαν εδώ και περιμένουν να δουλέψουν. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με το επιτελείο του και τον κύριο Μουγκουρούτσα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτήριο συνέδριο. Θα του δώσω αμέσως το λόγο για να μην καθυστερήσουμε άλλο. Παρακαλώ, κύριε Μουγκουρούζα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Γενική Γραμματέα της Ευρω... Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας για να σας παρουσιάσω τα βασικά αποτελέσματα του ελεγκτικού συνεδρίου, αυτή τη φορά όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, τις προηγούμενες εβδομάδες σας παρουσίασα τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, και τα θέματα διοίκησης. Ε, καταλήξαμε ότι το εκτιμόμενο επίπεδο σφάλματος είναι, είναι 0,6%. Ένα ποσό το οποίο διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια και είναι πολύ κάτω από το όριο το οποίο έχει ε, θέσει ε, το ελεγκτικό συνέδριο. Όσον αφορά τις 131 δράσεις, οι 84 ε, αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από αυτές που έγιναν στα πλαίσια του ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου. Είδαμε την διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων και κάποια σφάλματα στι δαπάνε προσωπικού που έκανε το Γραφείο για τα Ατομικά Δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ελληνικό Συνέδριο σε προηγούμενε διαδικασίε είχε ε, προτείνει να ληφθούν μέτρα ώστε να γίνεται περιοδικά ο έλεγχος ε, για την προσωπική κατάσταση των υπαλλήλων και να βελτιώσουμε και τα συστήματα ώστε να γίνεται επεξεργασία εγκαίρω όλων των πληροφοριών που θα μπορούσαν να έχουν υπάρχουν συνέπειε για τις ε, μισθού, τι συντάξει και τα οικογενειακά επιδόματα. Όσον αφορά την ετήσια έξεδεση του 2016, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ακόμα αυτέ οι αδυναμίες, επομένω επαναλαμβάνουμε τι συγκεκριμένε συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σα, κυρίε και κύριοι και θα... Ήθελα να σα πω ότι είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση ή να διασκεδάσω οποιαδήποτε αμφιβολία. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Πέρα από την ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, σήμερα θα εξετάσουμε και ε, τη συνέχεια, το follow-up της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περσινό έτος και έχουμε και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Η Γενική Γραμματεία έχει συστημικό ρόλο στην κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων. Ο Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Ιταλιάνα, έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά για μένα που είμαι εδώ για δεύτερη φορά υπό την ιδιότητά μου σαν Γενικό Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω το Ελεκτικό Συνέδριο για την ετήσια έκθεσή του και την παρουσίαση που έκανε ο κ. Μουγκουρούτσα. Επίση, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Τέλερ, για την πολύ καλή συνεργασία, την προετοιμασία τη ακροάσεω απαλλαγή. Ξυπακούεται ότι η Επιτροπή σα και το Συνέδριο παίζουν σωτικό ρόλο στην απαλλαγή του προπολογισμού και έχουμε κοινό όφελο εξασφαλίζοντα και το ότι ο προπολογισμό είναι αντικείμενο σωστού χειρισμού και ότι οδηγεί σε αυτά αποτελέσματα για του πολίτε. Τώρα από πλευρά συμμόρφωση το επίπεδο σφάλματο ήταν στα 3,8% το 2015 αντί 4,4% που ήταν το 2014. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, αλλά θα πρέπει να ξεκολουθούμε να επαγρυπνούμε και να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη που χειρίζονται το 80% του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Καλωσορίζουμε το ότι το Συνέδριο και το Κοινοβούλιο δίνουν όλο και μεγαλύτερη έμφαση στι επιδόσεις. Αυτό δείχνει, φαίνεται, στα κεφάλαια 3 στο κεφάλαιο 3 της ετησία εκθέσεως του Ελληνικού Συνεδρίου τον ορίζοντα 2020 δεν είναι μόνο σημαντικό να γίνεται σωστό ο χειρισμό των προγραμμάτων σύμφωνα με του κανόνε, αλλά θα πρέπει να αποδίδουν και να πετυχαίνουν του στόχου του. Και γι' αυτό η Επιτροπή Ευρωπαϊκή του κ. Γιούνκερ ε, τονίζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα. Εξετάζουμε κάθε πτυχή των ε, επιδόσεων του προπολογισμού, εστιαζόμενοι επί των αποτελεσμάτων βάσει τη κατάλληλη πρωτοβουλία και βελτιώνουμε τη διαχείριση τη επιδόση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορούμε να πετύχουμε του δικού στόχου και να διαθέτουμε του πόρου με τον αποτελεσματικό το δυνατό τρόπο. Το 2015 είναι το έτος που είναι το αντικείμενο της απαλλαγής. Να πω μερικά λόγια για τα επιτεύγματα του 2015. Βέβαια ήταν γεμάτο προβλήματα το έτος και πλευράς πολιτικής και πλευράς διαχείρισης του προπολογισμού. Αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές κρίσεις. Η προσφυγική κρίση είχε την ύψιστη προτεραιότητα. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις τρομοκρατικές επιθέσεις, την απαγόρευση των Ρώσων στις γεωρικές εξαγωγές, τη χρηματοστητική αστάθεια στην Ελλάδα, Αυτά ήταν απλώ μερικά από τα προβλήματα και αυτό ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκή Ενώσεω πιέστηκε. πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε ευελιξία για να διαθέσουμε τάχιστα του απαιτούμενου πόρου. Αυτή η εμπειρία απέδειξε ότι η μεγαλύτερη ευελιξία απαιτείται για να αντιμετωπίσουμε απροσδόκητε καταστάσει. Και γι' αυτό προτείναμε μεγαλύτερη ευελιξία στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Το 2015 ξεκίνησε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στατικές Επενδύσεις. Έδωσε πρόθεση, όθηση, μια κρίσιμη στιγμή για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Ταυτόχρονα η εμπροστοβαρής προσέγγιση για την απασχόληση των νέων έστειλε σημαντικό μήνυμα για την κοινή μας προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε τα παράδεκτα υψηλά επίπεδα ενεργείας των νέων. Το 2015 δεν αφορούσε μόνο την ανταπόκρισή μα στι κρίσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε και διάφορε φιλόδοξε στρατηγικέ για να πετύχει μακροπρόθεσμε πολιτικέ προτεραιότητε τη Επιτροπή Γιούνκερ. Εκεί συμπεριλαμβάνεται Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ανάστευση και την Ασφάλεια, στρατηγικέ για την ψηφιακή ενιαγορά, την Ενεργειακή Ένωση και την Ένωση τη Κεφαλαγορά, των Κεφαλαγορών μάλλον να πω μερικά πράγματα για το ρόλο τη γραμματεία, Γενική Γραμματεία εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2015 ήταν το πρώτο έτο εφαρμογή ε, των νέων μεθόδων εργασία τη Επιτροπή Juncker. Και αυτέ οι μέθοδοι έχουν σχεδιαστεί τόσο να εξασφαλίζουν στόχευση σωστά στι προτεραιότητε των Ευρωπαϊκών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην υπάρχει απομόνωση μεταξύ των διαφόρων τμήματων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να, να αποτελεσματικά του πόρου. Ε, η Γενική Γραμματεία έχει κεντρικό ρόλο στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτός ο ρόλος ε, ενισχύθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Γιούνκερ. Συντονίσαμε τις πολιτικές των υπηρεσιών μας ε, και για εκ μέρου του Προέδρου και εκ μέρου των Αντιπροέδρων. Υποστηρίζουμε και τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, διοργανώνοντα διάφορε ομάδε συγκεκριμένα θέματα, δίνουμε συμβουλές, ε, οργανώνουμε ενημερώσεις και ετοιμάζουμε διάφορα σχέδια κειμένων για βασικές πρωτοβουλίες. Αυτό είναι πέρα από τις παραδοσιακές ε, ευθύνε για την ομαλή λήψη αποφάσεων και για τη λειτουργία του θεσμού και σε θεσμικό και διαθεσμικό επίπεδο. Γι' αυτό ο Πρόεδρος αποφάσισε να ενισχύσει τη Γενική Γραμματεία με 80 θέσεις το 2015 το συζητήσαμε αυτό και πέρσι, το θέμα των στελεχών. Αυτές οι νέες θέσεις χρησιμοποιήθηκαν άριστα σε διάφορους τομείς. Φερρυπίν, ο Γενικός Γραμματέας συντόνισε και συντονίζει μέχρι σήμερα την ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση σε επίπεδο υπηρεσιών υπό την ηγεσία του Προέδρου και του πρώτου Αντιπρόεδρου. Ε, ο Γενικό Γραμματέα επίση έπαιξε ηγετικό ρόλο στο σχεδιασμό βασικών στρατηγικών πρωτοβουλειών, όπω Ενεργειακή Ένωση και Ψηφιακή Ενία Αγορά. Συνολικά ο Γενικό Γραμματέα συνέταξε πάνω από 70 ανακοινώσει και εκθέσεις ε, στα πλαίσια των στρατηγικών για την Επιτροπή Juncker και τι σχετικέ προτεραιότητε Juncker. Ο Γενικό Γραμματέα επίση συνέχισε να κατευθύνει τι εργασίε για τον απασχεδιασμό και την εφαρμογή και υλοποίηση του γενικού πλαισίου για την οικονομική διακυβέρνηση και το σχετικό ευρωπαϊκό εξάμεινο. Επίσης ανέπτυξε καλύτερο πακέτο για νομοθέτηση και έκανε προτάσεις για διοργανικές συμφωνίες, για καλύτερη νομοθέτηση και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων το 2016. Επίσης ξεκίνησε επικαιροποιημένη εκδοχή του Μητρώου Αδιαφανίας για να υποστηρίξει τις τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαφανή πολιτική. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε και πρόταση για υποχρεωτικό διοργανικό μητρό διαφανείας. Ο Γενικό Γραμματέας εξυγχρόνησε και απλούστευσε τη λήψη αποφάσεων μέσω του Decide που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα ψηφιοποίηση και λογισμικού. Τώρα για τη διαχείριση των επιδόσεων. Κάναμε σημαντικά βήματα για να σχέσουμε τη διαχείριση των επιδόσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Γενικός Γραμματέας το 2015 ξεκίνησε την, ε, τον εξυγχρονισμό του στρατηγικού σχεδιασμού και του προγραμματικού μας κύκλου, που είναι και το επίκεντρο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό συμπεριλαμβάνει σχεδιασμό, καθορισμό στόχων και υποβολή εκθέσεων. Μέσω της μεταρρυθμίσεως προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την ε, ποιότητα, να μειώσουμε τον αριθμό των στόχων και των δικτών, βοηθώντας αυτό να εστιαζόμεθα επί των σημαντικών ζητημάτων. Ακρογωνιός λήθο του νέου συστήματος που ανακοίνωσα πέρσι είναι ο πολιετής ε, σχεδιασμός που κατατίθεται από κάθε γενικό διευθυντή. Αντί να δημιουργούμε νέους στόχους και δείκτες κάθε χρόνο, όλες οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εκπονήσει ε, σταθερά σχέδια για το 2016-2020 για αυτή την περίοδο ε, για να υπάρχει και μια συνέπεια μεταξύ υπηρεσιών. Αφετηρία του σχεδιασμού είναι οι 10 πολιτικές προτεραιότητες Α, είμαι πολύ γρήγορο. Και εγώ έλεγα ότι πάω. εντάξει, θα πάω πιο σιγά. πάω Αφετηρία λοιπόν για το σχεδιασμό είναι οι 10 πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ και εκφράζονται σαν γενικοί στόχοι. Συνοδεύονται από δείκτες συνεπιών για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο. Και αυτοί οι δείκτες συνεπιών συμπεριλαμβάνουν όλους τους στόχους ε, των κατηγοριών για την ε, Ευρώπη του 2020. Ε, εκεί δείχνουμε πώς ταιριάζουν προτεραιότητες με τη στρατηγική για ανάπτυξη και απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο στρατηγικό σχεδιασμό, οι γενικοί διευθυντές εξηγούν το πώς οι δραστηριότητέ του συμβάλλουν στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπή αυτό επιτυγχάνεται υπό τη μορφή συγκεκριμένων στόχων, αναπερίπτωση και κατάλληλους δείκτες αποτελεσμάτων. Εντός αυτού του πλαισίου λοιπόν, του στρατηγικού σχεδιασμού, το ετήσιο διαχειριστικό σχέδιο χρησιμοποιείται για να εξηγήσει το πώς τα αποτελέσματα του έτους συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων. Οι γενικοί διευθυντές λοιπόν θα ενημερώνουν επί των νέων στόχων και δικτών για πρώτη φορά στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, έκθεση δραστηριοτήτων ε, φέτος. Θα γίνει για πρώτη φορά αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι το νέο σύστημα είναι σημαντικότατο βήμα πρόοδου για διαχείριση των επιδόσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φρονούμε ότι είναι ένα βήμα που συγκρίνεται ευνοϊκά με τα εφιστάμενα συστήματα σε άλλους δημόσιους φορείς. Πράγματι. Τίθενται οι πολιτικέ προτεραιότητε, οι κατάλληλε και για την Ευρώπη του 2020 και καθώς αφορά τις 10 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Όλα αυτά μπαίνουν στο επίκεντρο των προσπαθειών μα. Αυτό το νέο σύστημα έχει πραγματικά αποτελέσματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε του πόρου μα. Το 2016 για πρώτη φορά θεσπίσαμε μια νέα μεθοδολογία για την κατανομή του προσωπικού μεταξύ των τμήματων μας. Αυτό συμβάλλει στον καθορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και είναι βασικό κριτήριο αυτό για τις αποφάσεις που λαμβάνονται για τη διανομή του προσωπικού. Ε, πάμε τώρα στην ετήσια διαχείριση και την έκθεση των επιδόσεων. Πέρσι παρουσίασα την έκθεση εξολόγηση του 2014 βάσει του άρθρου 380 ε, σε αυτή την Επιτροπή και ανακοίνωσα ότι το 2015 θα κινηθούμε προς πιο ολοκληρωμένη έκθεση όσον αφορά οικονομικά. Σύμφωνα με τις συστάσεις και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Συστάσεις που έγιναν περίπου δύο χρόνια πριν. Αυτό, αυτή η νέα έκθεση επιδόσεων και διαχείρισης συγκεράζει δύο πρώτες εκθέσεις. Την έκθεση αξιολόγησης, δυνάμει του άρθρου 380 που ανέφερα πριν, και την πρώην συναπτική έκθεση για τη διαχείριση των επιτεγμάτων μάλλον τα επιτέματα των διαχειρήσεων. Έτσι έχουμε καλύτερη εικόνα των επιδόσεων. Καλύπτουμε και το πώς αποδίδουν τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πώς χειρίστηκε και εξετέλεσε τον προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αντιπρόεδρος κυρία Γεωργίευα παρουσίασε την έκθεση αυτή σε εσά τον περασμένο Οκτώβριο. Η μορφή της εκθέσεως άλλαξε. Όμω εξακολουθούμε να ακολουθούμε τι πολύ χρήσιμε συστάσει του Ευρωκοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη δομή αυτή και το περιεχόμενό τη. Παραδείγματο χάρη, παρουσιάζουμε πληροφορίε κατά κατηγορίε του προπολογισμού, εξηγούμε πώ συμβάλλει ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την επιτύχηση των στόχων τη Ευρώπη 2020 και δίνουμε παραδείγματα τη τη αξία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η δυνατότητα τα ερευνητικά προγράμματα να καλύπτουν πανευρωπαϊκά προβλήματα. Υποσχέθηκα πέρσι, σας υποσχέθηκα ότι θα ελπίζαμε να σας δώσουμε πληρέστερη εικόνα όσον αφορά την έκθεση του 2015 για τις επιδόσεις κάποιων βασικών μας προγραμμάτων για τις προηγούμενες περιόδους. Πράγματι, αν δείτε την έκθεση, συνοψίζει τα αποτελέσματα διαφόρων νέων εκτονιστέρων αξιολογήσεων. Να σας δώσω ακροθυγώς κάποια παραδείγματα. Πρώτον, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, το ερευνητικό, είχε έμεσα οικονομικά αποτελέσματα της κατηγορίας των 20 δισεκατομμύριων ευρώ ετησίως. Υποστήριξε 11 ανθρώπους που πήραν το βραβείο Νόμπελ. Μετά επενδύσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης δημιούργησαν 825.000 θέσεις απασχόλησης και βοήθησαν πάνω από 20.000 ε, επιχειρήσεις. Τέλος, αυτές οι αξιολογήσεις αποδεικνύουν ότι οι φοιτητές που μελέτησαν στην Αλοδαπή χάρη στο Εράσμους, στο πρόγραμμα Εράσμους, αύξησαν την δυνατότητα απασχόλησής τους σε σχέση με φοιτητές που δεν είχαν μετακινηθεί κατά 45%. Αυτά ήταν παραδείγματα για την πρώτερη προγραμματική περίοδο. Είναι πολύ πρόημο τώρα να σα ενημερώσω λεπτομερώ για την τρέχουσα περίοδο. Κάποιε αρχικέ ενδείξει όμω ήδη δείχνουν θετικέ ε, τάσει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανακοίνωσα πέρσι ότι θα αυξήσουμε την υποβολή εκθέσεων και την ενημέρωση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων και στην ετήσια έκθεση διαχείρισης ε, ε, και αποτελεσμάτων μπορούμε να πούμε ότι 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις και διάφορα σχετικά προγράμματα υποστηρίχθηκαν από αυτό το ταμείο, το ταμείο Γιούνκερ όπως αποκαλείται, από τον Μάιο πέρσι. Έκτοτε δημοσιεύσαμε τρεις αξιολογήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ένας εξωτερικός ελεγκτικός φορέας Όλες οι εκθέσεις αμπόρισμα είχαν ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στατηγικές Επενδύσεις πέτυχε, πρόθεσε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και κινητοποίησε και το ιδιωτικό κεφάλαιο. Ε, αυτό στηρίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, τον διπλασιασμό και της διάρκειας και του, των οικονομικών δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στατικές Επενδύσεις και ελπίζουμε ότι αυτές οι προτάσεις τελικά θα στηριχθούν και μάλιστα γρήγορα. Άλλη μια υπόσχεση που έκανα πέρσι ότι θα σε ενημερώσω για τα αποτελέσματα μόχλευσης μέσω ε, της πρωτοβουλίας μας για τα διάφορα προγράμματα που είναι πρόδομος του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, Στρατηγικών Επενδύσεων και εξωτερική αξιολόγηση είδε ότι το, είχαμε μόχλευση 12,9 της τάξης του 12,9 υψηλότερο από αυτό που είχαμε ε, υποβάλει ως αποτέλεσμα πέρσι. Και για τα δύο παραδείγματα βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες ε, στα συγκεκριμένα κείμενα των ειδικών αυτών εκθέσεων. Υπάρχει και κάτι γενικότερο που θα ήθελα να τονίσω για την ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων και διαχείρισης και αποτελεσμάτων. Είναι είσοδος, αν θέλετε, σε λεπτομερέστερες πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις προγραμμάτων που προσαρτώνται κάθε χρόνο στο σχέδιο προπολογισμού. Επίση, πληροφορίε που περιέχονται στι εκθέσει αξιολογήσεως και στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Και, ενημερω... και δείχνουμε λεπτομέρω ποια είναι η πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων Ευρώπη 2020 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τέλο, εκπονούμε επικαιροποίηση όσον αφορά την πρόοδο, όσον αφορά τι 10 προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, φυσικά, πάντα προσπαθούμε να βελτιώσουμε το σύστημα ενημέρωσης και συντάξει εκθέσεων και χαιρόμαστε που του χρόνου το ελεκτικό συνέδριο θα συγκεντρωθεί επί των εκθέσεων επιδόσεων στο κεφάλαιο 3 της ετήσιας εκθέσεως και προσβλέπουμε σε συζητήσεις με το συνέδριο και στην ε, αντίστοιχη τέτοια συνεδρίαση του επόμενου έτους. Κλείνοντας λοιπόν, κυρία Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη, παρόντα μέλη, θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπα και πέρσι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νοοτροπία επιδόσεων, αλλά αυτό χρειάζεται χρόνο. Επίση, είναι κοινή ευθύνη αυτή. Έδωσα διάφορα παραδείγματα σήμερα για το πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα διάφορα θέματα και ενημερώνουμε και συντάσσουμε χθε τι επιδόσει. Θέλουμε υποστήριξη από το Συμβούλιο και, την, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεκτικό Συνέδριο. Είναι κρισίμου σημασία, όπω είναι στον τομέα τη συμμόρφωση και των οικονομικών ελέγχων. Γι' αυτό χαίρομαι που ξεκινούμε τη συνεργασία μα μέσω τη ομάδα εμπειρογνωμόνων για, τον, για την κατάρτιση προπολογισμού βάση επιδόσεων. Πρέπει να συνεννοούμεθα όσον αφορά το τι νοούμε με επιδόσει και πώ προσμετράτε αυτό και αυτό είναι βασικό στοιχείο για την πρόοδο στον τομέα. Συλλέγουμε πληροφορίε. Αυτέ θα τροφοδοτήσουν τον προβληματισμό μα και εργασίε για τον προπολογισμό που θα έχει στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα και κάποια τα συμπεράσματα και πορίσματα των εργασιών αυτών ενέπνευσαν τις προτάσεις μας για την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και πιο συγκεκριμένα την ανάγκη για περαιτέρω απλούστευση και ευελιξία του προϋπολογισμού. Όμως, νομίζω ότι η δυνατότητα για πραγματική πρόοδο θα έρθει με τις προτάσεις για τη νέα γενιά των προγραμμάτων, για, το, για τη νέο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και ενδιάμεση αξιολόγηση δείχνει αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των εστώτος έτους. Τέλος λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει κάθε προσπάθεια να αποβάλει προτάσεις την κατάλληλη στιγμή που θα είναι φιλόδοξες και θα επιφέρουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η συγητή της Επιτροπής μας είναι ο κύριος Τσέλερ και του δίνω αμέσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχά να ζητήσω συγγνώμη για την αργοπορία μου. Αυτά συμβαίνουν όταν πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα και στην προκειμένη περίπτωση μια προετοιμασία για αποστολή τη επιτροπή ανάπτυξη. Έπρεπε να συζητηθούν κάποια θέματα για αυτή την αντιπροσωπεία. Συγγνώμη λοιπόν. Γι' αυτό άργησα. Ευχαριστώ πολύ και τους ε, κυρίους, ε, τον κύριο Μουγκουρούζα από το Ελεκτικό Συνέδριο και τον Γενικό Γραμματέα κύριο Ιταλιάνε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λεπτομερέστατη παρουσίαση που έκαναν και για την καλή συνεργασία που έχουν δείξει μέχρι τώρα. Τα ποσοστά ασφάλματος είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με τις διοικητικές δαπάνες. Ο κύριος Μουγκουρούζα το ανέφερε. Είναι πολύ σωστό αυτό, είναι και πολύ σημαντικό να λειτουργούμε με τρόπο υποδειγματικό. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο επίκεντρο αυτής της διεργασίας. Είναι λοιπόν κάτι που μας χαροποιεί. Μετά, έχω κάποιες ερωτήσεις, κάποιες παρατηρήσεις, ωστόσο όχι για το ΕΦΣΥ. Αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλο σημείο της συνεδρίασης, αλλά για τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2016 έκανε μια πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας συγκεκριμένα χαιρετίζουν την πρόταση αυτή για επικαιροποίηση των κανόνων σε σχέση με την διάθεση των κονδυλίων. Ωστόσο, βλέπουμε έναν κίνδυνο οι πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις να καταλήξουν να είναι αντιπαραγωγικές. Η τελευταία ε, εκδοχή του κανονισμού τέθησε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016 και θα ισχύει μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ανακοινώνει ε, θεμελιώδεις αλλαγές στην πρότασή της, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Ε, ακόμα και αν εγκριθεί λοιπόν ο νέος κανονισμός μέχρι το Σεπτέμβριο, θεωρώ πως είναι προβληματική η εφαρμογή του ακριβώς λόγω του διοικητικού άχθους, λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας στην εφαρμογή της. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν μέσα σε ένα ελάχιστο διάστημα μερικών μηνών να μπορούν να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές. Επίσης δεν βλέπω ε, κάποια εκτίμηση αντικτύπου στην πρόταση και θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί. Τώρα σε σχέση με τις επιδόσεις. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας ε, υποστηρίζει έναν προϋπολογισμό καταρτισμένο βάσει επιδόσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο ε, αυτό, αλλά η αξιολόγηση. Είναι, πιστεύουμε, η βάση για όλες τις επόμενες αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν και πολιτικές επιπτώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η αξιολόγηση πρέπει να ληφθεί υπόψη το συντομότερο δυνατό, διότι διαφορετικά θα δημιουργηθούν προβλήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα πώς εσείς ε, θεωρείτε πως μπορούμε να δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτήν την αξιολόγηση ε, μέσω των εκθέσεων και πώς θα δώσουμε στο ηλεκτρικό συνέδριο αρκετό χρόνο έτσι ώστε να διεξάγει την αξιολογηση μεσω των εκθεσεων και πως θα δωσουμε στο ηλεκτρικο αυτή. Τώρα, ε, ο κώδικας δεοντολογίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Εδώ και πολλά χρόνια ζητούμε μια ε, επανεξέταση των κανόνων και έναν σαφέστερο ορισμό της σύγκρουση συμφερόντων. Ζητάμε επίσης για πάρα πολύ καιρό συγκεκριμένα κριτήρια για το χρονοδιάγραμμα, για, την για το διάστημα απασχόλησης και ζητούμε ένα χρονικό διάστημα τριών ετών ο προηγούμενος ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος ε, Μπαρόζο, όπως γνωρίζετε, έχει αναλάβει ένα νέο πόστο και η ακρόαση της ε, κυρίας Αγγεωργίρβα τον Οκτώβριο έθεσε ορισμένα ερωτήματα. ακριβώς λόγω της ε, θέσης της ως Επίτροπο Προϋπολογισμού. Άλλαξαν λοιπόν ορισμένα πόστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, ακριβώς λόγω όλων αυτών των αλλαγών, λόγω αυτών των εξελίξεων πιστεύουμε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επανεξέταση της κατάστασης. Ο πρόεδρος Γιούνκερ στο τέλος του περασμένου έτους μας ε, είπε ότι θέλει να ε, παρατείνει την ε, θητεία του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό όμως πρέπει να το κοιτάξουμε. Τώρα, εγώ έχω μια ερώτηση και για τον αριθμό των απασχολούμενων στη Γενική Γραμματεία. Βλέπω τις εξελίξεις στον αριθμό των υπαλλήλων και νομίζω πως ε, παρατηρώ πως υπάρχει μεν μεγαλύτερη απασχόληση, λιγότερες πρωτοβουλίες ε, πολιτικού χαρακτήρα όμως. Αυτό βέβαια ήταν και μία πρωτοβουλία του Προέδρου της Κομισιόν, οποίος ήθελε να μετριάσει λίγο αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια συμφωνία που μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις γραπτές απαντήσεις που μας δώσατε, να σας ευχαριστήσω καταρχάς Έχω όμως και κάποιες ερωτήσεις για το σημείο 3 για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πόσες φορές συναντήθηκε το 2015 Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μετά, Task Force, σημείο 6, ε, δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει κάποια απάντηση από το διοικητικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο των δημοψηφισμάτων. Μετά, ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσαμε και τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει για να αποφύγουμε τον Brexit. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά την ερώτηση, το σημείο 21, εκτίμηση αντικτύπου. Ε, δημοσιεύτηκε πρόσφατα μία μελέτη από το Ινστιτούτο Εκτίμησης Αντικτύπου και Επιστημονικής Αξιολόγησης Πολιτικής ε, για το θέμα της καλύτερης νομοθεσίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν υποβληθεί πολλές νομοθετικές προτάσεις χωρίς ε, πρώτερη εκτίμηση αντικτύπου ή χωρίς πλήρη εκτίμηση αντικτύπου. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω γιατί. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον συγγετή τον κύριο Τσέλερ για την ε, αγαστή συνεργασία καταρχάς και για τις πολύ καλές ερωτήσεις που μου έθεσε. Θα κάνω μια απόπειρα να απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό που πρότεινε εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρώ ότι είναι μια συνεκτική πρόταση για απλούστευση, όχι μόνο όσον αφορά τις αλλαγές στο δημοσιονομικό κανονισμό, αλλά είναι και σε σχέση με την πρόταση Omnibus, όπως αποκαλείται, για τις αντίστοιχες αλλαγές ε, στην ομοθεσία. Αρκετές από αυτές τις προτάσεις απλούστευσης ήδη αποτελούσαν τμήμα της αρχικής πρότασης ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο αυτή τη στιγμή ισχύει, και ε, είναι και κάτι το οποίο ε, λήφθη υπόψη στη διαπραγμάτευση για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, κατά μία έννοια λοιπόν ε, πολλές από τις προτάσεις δεν ε, αποτελούν κάτι καινούριο. Προσπαθήσαμε όμως να έχουμε μία συνεκτική πρόταση σε αυτή την περίπτωση. Βεβαίως αν αλλάζει πολύ συχνά ο δημοσιονομικός κανονισμός αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες και στους δικαιούχους αλλά και στις ε, διοικήσεις. Δεν θα μπορούν να σεβαστούν εύκολα τους κανόνες. Ε, αφετέρου θεωρώ ότι η απλούστευση είναι κάτι ε, πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν ε, απτά παραδείγματα στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 όπου ποτέ δεν αρκεί η απλούστευση και ρωτήσατε επίσης γιατί δεν έγινε αξιολόγηση επιπτώσεων για ε, την ε, πρόταση αυτή. Από τη μια μεριά, πολλά από αυτά τα στοιχεία της απλούστευσης ήδη περιλαμβάνονται στις αρχικές προτάσεις ε, και όταν προτάθηκαν ως τμήμα του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, επομένως καλύφθηκαν και από τις αξιολογίες επιπτώσεων που έγιναν τότε. Δεύτερον, ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών. Δεν είναι πολύ εύκολο λοιπόν να γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων ε, για το περιβάλλον, παραδείγματο χάρη, ε, του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το διοικητικό άχθος, ε, παραδείγματος χάρη, του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό αξιολογήθηκε σε έγγραφα τα οποία συνοδεύουν τις προτάσεις μας. Τέλος, υπήρχε και μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης πριν την υποβολή της πρότασης. Στη συνέχεια ρωτήσατε για τις επιδόσεις και την ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων και τη σχέση με την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εορτή. Υπάρχει μια εκ των προτέρων αξιολόγηση υπό τη μορφή αξιολόγηση επιπτώσεων, αλλά η εκ των υστέρων αξιολόγηση πρέπει να γίνει όταν θα έχουν οριστικοποιηθεί τα πάντα. Υπάρχουν καθυστερήσει, καταρτίζονται προτάσεις, εγκρίνονται στη συνέχεια και εφαρμόζονται. Πάντα ε, τίθεται θέμα και χρονικής διάρκειας ε, μεταξύ τη αρχική αξιολόγηση και τη υποβολή νέων προτάσεων επειδή δραστηριοποιούμαστε σε ένα τομέα που είναι σχετικά σταθερό, αυτό δεν έχει και τόσο σημασία, διότι το πλαίσιο για τα προγράμματα μπορεί σίγουρα να βελτιωθεί και αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν πιο περίπλοκα όμως όταν κινούμαστε προς νέους τομείς. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε ενδιάμεσες αξιολογήσεις, ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση. Προσπαθούμε να θέσουμε στόχους όσο μπορούμε στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και να επικαιροποιήσουμε πράγματα. Είναι ένας πιο απλός τρόπος να προσεγγίσουμε ε, τα όσα προβλέπει η αξιολόγηση. Τέλος, όσον αφορά την ε, έκθεση για τις επιδόσεις, η έκθεση η οποία είναι τμήμα της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης συνήθως δημοσιευόταν νωρίτερα. Αυτό όμω ε, είναι τρόπον την το τίμημα ε, που πληρώνουμε ε, για λόγους συνέπειας. Η συνέπεια είναι πάρα πολύ σημαντική και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Ελεκτικό Συνέδριο και υπήρχαν συστάσεις για τον εξορθολογισμό πριν από ένα-δύο χρόνια. Μετά ρωτήσατε για τον κώδικα διοντολογίας. Ο πρόεδρος Γιούνκερ για το θέμα αυτό ανακοίνωσε στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θέλει να αλλάξει ο κώδικας διοντολογίας σε δύο πτυχές κυρίως. Η πρώτη είναι για το θέμα της εκλογικής άδειας και η δεύτερη είναι για τη διάρκεια της λεγόμενης περίοδου cooling off για τα πρώην μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο πρόεδρος ε, διαβουλεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως πρέπει να κάνει βάσει και τις συμφωνίες πτυχές. Κατόπιν είχαμε μια ερώτηση για το προσωπικό και την πιθανή αντίφαση που υπάρχει μεταξύ ανάθεσης περισσότερου προσωπικού, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λιγότερες πρωτοβουλίες. Όπως σας είπα ήδη, πολλές από τις νέες πρωτοβουλίες καταρτίστηκαν ε, με την ευθύνη των αντιπροέδρων και η Γενική Γραμματεία ε, εξυπηρετεί τους αντιπροέδρους, επομένως αυτό το επιπλέον προσωπικό χρησιμοποιήθηκε για να βοηθήσει τους αντιπροέδρους για τις νέες πρωτοβουλίες. Παρά το γεγονό ότι ο συνολικό αριθμό πρωτοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μικρότερο. Ε, είναι θέμα ε, σχετική κατανομή προσωπικού εντό των υπηρεσιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι προσθήκη προσωπικού. Ερωτήσατε για τι επισκέψει προ τα Εθνικά Κοινοβούλια των Επιτρόπων. Ε, τα στοιχεία τα οποία έχω εγώ ε, λένε ότι το 2015 είχαμε πάνω από 200 επισκέψεις. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι λαμβάνουμε όλο ένα και περισσότερες γνωμοδοτήσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, είτε στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας κίτρινης κάρτας, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει πλειοψηφία για την υποβολή κίτρινης κάρτας ε, και τη σχετική πρωτοβουλία, απαντούμε σε όλα τα κοινοβούλια ξεχωριστά και ο αριθμός αυτός ανέβηκε το 2016 και λάβαμε πάνω από 600 γνωμοδοτήσεις από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τέλος, ε, ρωτήσατε για την Task Force ε, για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ρωτήσατε κατά πόσον η Task Force αυτή ήταν επιτυχής. Ε, νομίζω ότι αυτό δείχνει ε, τα όρια της ε, διαχείρισης βάσει επιδόσεων. Δεν θα έλεγα ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχέση με το ρόλο της συγκεκριμένη Task Force, αλλά πρέπει να πω ότι ήταν αρκετά χρήσιμη γιατί μπόρεσε να προετοιμάσει τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συμφωνία στην οποία κατέληξαν με το Ηνωμένο Βασίλειο για το δημοψήφισμα για να δούνε τα όρια αυτών που μπορούμε να παραχωρήσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του παρόντος πλαισίου. Και αν αυτό αποτελεί μέτρο επιτυχία, νομίζω ότι η Task Force ήταν ιδιαίτερα επιτυχη. Αναφερθήκατε επίση στο ρόλο τη Task Force για την εκστρατεία για το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να υπενθυμίσω ότι υπήρχε πολύ συγκεκριμένο αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου να μην συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την ε, εκστρατεία. Και φυσικά σεβόμαστε τι επιλογέ ε, του συγκεκριμένου κράτου μέλου. Τέλος. Ρωτήσατε για το Brexit. Η Task Force για το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου εντωμεταξύ διαλύθηκε και τώρα υπάρχει μια Task Force για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, που είναι μια πολύ μεγαλύτερη Task Force. Προεδρεύει ο Μισελ Μπαχνιέ Και το πρώτο σημαντικό καθήκον αυτή τη ομάδα ειδικών καθηκόντων είναι να δει ποια είναι η επιθυμία, να σεβαστεί μάλιστα και την επιθυμία των ε, ε, πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτή η επιθυμία να ε, εκπληρωθεί με συγκεκριμένο σωστό τρόπο, να δούμε ποιες μπορούμε να έχουμε, τι μπορούμε να έχουμε ως μελλοντικέ σχέσεις και πώς μπορούμε να έχουμε μια ομαλή μετάβαση στο μελλοντικό πλαίσιο. Και βεβαίω η Task Force έχει ω στόχο να επιτύχει αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να εκτιμούμε το χιούμορ σα Το συμμεριζόμαστε. Αλλά νομίζω πω ήταν λάθο να μην συμμετέχουμε και εμεί σε αυτό το δημοψήφισμα και να μην επιτρέψουμε στου απερχόμενου επιτρόπου να παραθέσουν κάποια γεγονότα κάποια στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες. Νομίζω πως ε, δεν υπήρχε παρκής πληροφόρηση. Ε, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Λιμπεράτσκι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, να πω πως έχω κάπως ανάμεικτα αισθήματα. Από τη μία φαίνεται πως όλα βαίνουν καλώς, δεν υπάρχει μεγάλο ποσοστό σφάλματος, από την άλλη όμως έχω την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει και τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Πως υπάρχει μια παθητικότητα και δεν βλέπω αυτήν την ηγετική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα στο θέμα του Brexit. Δεν είδα κάποια ανάληψη πρωτοβουλίας, είδα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, άπραγη σχεδόν. Όμως, να μείνω στο θέμα μας, την απαλλαγή. Ακούσαμε πως πρέπει να είμαστε βασισμένοι σε αποτελέσματα. Ο κύριος Τσέλερ είπε αρκετά, τα οποία πιστεύω δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρειάζεται να ακούσει αυτά, αυτές τις φωνές. Δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει βέβαια επιθυμία να γίνει απλοποίηση των κανόνων, όμως στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Οι κανόνες γίνονται όλο και πιο δύσκολοι, η σύγχυση μεγαλώνει. Μετά, ε, σε ό,τι αφορά τον κώδικα διοντολογίας. Νομίζω πως έχει πληγεί η φήμη μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται ανακοινώσει χωρίς όμως να γίνονται πράξεις. Πολλές φορές μάλιστα ακούω σχόλια ότι για παράδειγμα όποιο εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω επίτροπο, για παράδειγμα αυτό χρησιμοποιείται μόνο ως εφαλτήριο για κάποια ακόμα καλύτερη θέση. Και πρέπει να τοποθετηθούμε, πρέπει να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε η διοίκηση και εδώ μια παράκληση από μένα να μας ενημερώνει. Και η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το προσωπικό υπάλληλο να ασχολείται πραγματικά με τις αρμοδιότητές τους. Διότι η πραγματικότητα διαφέρει και βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζει στον Άρη. Δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Δεν βλέπει τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με συγχωρείτε για τη σκληρή διατύπωση, όμως πιστεύω πως έχει έρθει η ώρα να το πούμε έξω από τα δόντια. Για να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Τώρα, ε, σχέδιο Juncker. Είναι ένα πρόγραμμα με 10 σαφείς Βλέπουμε όμως ότι και σε αυτή την περίπτωση ακούγονται κατηγορίες εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι για παράδειγμα δεν υπάρχει γεωγραφική ισορροπία στο σχέδιο Juncker, δεν υπάρχουν πληροφορίες ε, για την προσβασιμότητα στα κονδύλια, στη χρηματοδότηση. Τι είναι όμως αυτό το σχέδιο Juncker, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει μια γενικότητα, οι πολίτες δεν είναι παρκώς ενημερωμένοι, Πολλές φορές βέβαια στην πολιτική έτσι είναι τα πράγματα και σίγουρα δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις, υπάρχουν χαζές απαντήσεις. Τώρα, μια ερώτηση προς τον κύριο Γενικό Γραμματέα. Ή μάλλον και ένα σχόλιο μαζί. Η δική μου πολιτική ομάδα αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση να δημιουργεί θετικά ερεθίσματα, να ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εικόνα της με τις πράξεις της. Σε αυτή την έκθεση δεν βλέπουμε αυτό το ηγετικό πνεύμα καθόλου. Αυτά ε, ήταν τα όσα ήθελα να πω εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας. Ε, και τώρα, σε ό,τι αφορά τις γραπτές απαντήσεις, ο κύριος Τσέλερ ήδη αναφέρθηκε με πολλές λεπτομέρειες αυτό, γι' αυτό δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ε, το μόνο που έχω να πω είναι μια τελευταία παράκληση για περισσότερη σαφήνεια, περισσότερη ουσία, περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη ανάληψη πρωτοβουλίας. Αυτό πιστεύω θα έκανε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ε, να κάνει τη διαφορά και να αλλάξει την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που μας λείπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, για να απαντήσει όμως ο Γενικός Γραμματέας, σας παρακαλώ να είστε σύντομοι όλοι. Ε, το λόγο έχει η κυρία Λαμπάγιοβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ιταλιάνερ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ για τις γραπτές απαντήσεις που μας δώσατε. Να ξεκινήσω από κάτι ωραίο, κάτι light η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνει προσπάθειε σε πρώτου διορισμού, ε, είπατε. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Και έχουν διοριστεί ε, νέα στελέχη μεσαίου επίπεδου. Έχουμε φτάσει στο 48% το 2016. Έχουμε μεγάλη αύξηση στην τάση. Σας διαβεβαιώ ότι ακόμα μετά την αναχώρηση της Αντιπροέδρου Γεωργίευα θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για την ε, ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων το 2018. Ας πάμε σε κάτι πιο επίκαιρο. Ακούσαμε και από άλλους συναδέλφους η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προβλήματα και εξωτερικά και εσωτερικά που ίσως επηρεάζουν και τη μελλοντική της ύπαρξη. Αυτό δεν είναι πολύ καλή συγκυρία για την 60η επέτειο. Χρειάζεται προβληματισμό. Να δούμε ποια είναι η νέα κατάσταση. Ποια είναι η κατανομή των διαφόρων ευθυνών σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, εθνικό επίπεδο περιφερειακό. Πρέπει να προσαρμοστούν οι δυστυχίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση για να επιληθούν τα παρόντα προβλήματα. Να αποφύγουμε ε, να αποφύγουμε ανάμειξη των διαφόρων δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Να δώσουμε πραγματική προστιθέμενη αξία όσον αφορά τι εργασίε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω για όλα τα κράτη-μέλη. Πολλέ τρέχουσε δραστηριότητε απομονώνονται σε συγκεκριμένε γενικέ διευθύνσει. Δεν υπάρχει επαφή με τι άλλε γενικέ διευθύνσει. Δεν υπάρχει κατάλληλη συνεργασία και συμπληρωματικότητα. Άρα χρειάζεται συνεργασία μεταξύ γενικών διευθύνσεων. Αυτό θα βοηθήσει στη σωστή επίλυση των προβλημάτων. Μετά από δύο χρόνια, πώ αξιολογείτε την νέα οργάνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που βασίζεται σε συνεργασία μεταξύ των αντιπροέδρων και οριζόντια προσέγγιση για κάποιε δραστηριότητε. Πώ το βλέπετε, Χρειάζεται η αρχή τη επικουρικότητα εφαρμόζεται. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινείται μόνο σε δραστηριότητε που δίνουν συγκεκριμένη ε, προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην αναμειγνύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εθνικέ δραστηριότητε. Έχετε γενικού κανόνε για τι γενικέ δραστηριότητε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Εγώ ήμουν υπεύθυνη για την απαλλαγή του 2014. Αλλά δεν ξέρω ποια συνέχεια δόθηκε όσον αφορά το δεντολογικό κώδικα για επιτρόπους το αναφέρατε εσείς, το αναφέρε και ο εισηγητής ο κ. Τσέλερ, αλλά δεν βλέπω κάτι συγκεκριμένο. Θα έπρεπε ίσω ε, βάσει τη γενική αντίληψη υπάρχει για το εντολικό κώδικα να επιφέρει κάποιε βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω ο κ. Τζέλερ, και εγώ τονίζω ότι υπάρχει έλλειψη αξιολογήσεω αντικτύπου. Κάτι που μου χρειαζόμαστε. Εγώ επεξεργάζομαι κάποια θέματα προσωπικά και δεν μου αρέσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αναθωρήσει οδηγιών χωρίς να περιμένει την υλοποίηση και εφαρμογή των οδηγιών επιβολής και να μην περιμένει για εκθέσεις αντιχτύπου. Ξέρετε σε τι αναφέρομαι. Χρειαζόμαστε χρόνο για όλα αυτά, αλλά σας ευχαριστώ για τις ε, εκ των προτέρων για τις αντιδράσεις αυτά. Ευχαριστώ, συνάδελφε Φλάνναγκαν, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, εκπλήσω με κάπως έχοντας ακούσει αυτά που είπατε για το Brexit και τον αντίκτυπο που είχε η ομάδα κρούσης, η Task Force. Τι είπατε, ε, τι να κάνουμε, σηκώστε χέρια στον αέρα. Καλό είναι τα βλέπουμε κάπως αστεία, ε, θα λυνόταν πολλά προβλήματα. Αυτό που θα λύσει το πρόβλημα η απομάκρυνση από την πραγματικότητα ο, θεσμός στον οποίο εργαζόστε έπαιξε σημαντικό ρόλο για το Brexit. Δεν συνέβη από μόνο του το Brexit, απομονωμένα. Τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Συνέβη το Brexit λόγω δυσαρέσκειας ε, για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Μπορεί να άπειρα εργαστήρια και άπειρα φόρα, αλλά όσο το κοινό της Ευρωπαϊκής Ενώσης ε, πιστεύει ότι κάτι τρέχει εκεί, σίγουρα ο κόσμος θα απομακρυνθεί από τα όνειρά σας της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Ένα παράδειγμα. Το ανέφερε και ο συνάδελφος ο κ. Λιμπεράτσκι. Ο κ. Μπαρόσο και οι πρώτεροι επίτροποι. Υπήρχε η αντίληψη ότι η δουλειά που έκαναν ήταν απλώ να χρησιμοποιούν τη θέση του για εφαλτήριο για μεγαλύτερα πράγματα. Αυτή είναι η αντίληψη του κόσμου. Έτσι το βλέπουν. Ο μόνο τρόπο να το αλλάξει κανεί αυτό είναι να σκοτώσουν αυτή την αντίληψη εξασφαλίζοντα ότι οι συγκρούσει συμφέρονται. Και δεν έπρεπε να συμβούν εξ αρχή οι συγκρούσει συμφερόντων. Ένα άλλο λόγο για τον οποίο συνέβη το Brexit και θα συμβούν και άλλα τέτοια γεγονότα είναι διότι η απόφαση κυριάρχων κρατών και τη Βρετανία και η Βρετανία θέλει να είναι κυριαρχό κράτο απορρίπτονται οι αποφάσει των κυριαρχών κρατών. Αν δεν είναι αρεστή η απόφαση κυρίαρχου κράτου, λέτε Α, έκανε λάθο η χώρα. Το είπε και η πρόεδρο. Όπω ε, το έζησε και ο λαό τη Ιρλανδία. Όταν δεν ψήφισε όπω ήθελαν για τη Λισαβόνα και την Νίκαια, του είπαν Κοιτάξτε, κάνετε λάθο. Αν συμφωνείτε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συμφωνεί κανεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται έξυπνο, μορφωμένο, ότι ξέρει τι τρέχει και αν διαφωνεί κανεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι κάνει λάθο. Δεν ξέρω. Τον φασισμό, είδατε τη λέξη φασισμό, τον ορισμό του φασισμού. Κοιτάξτε ποια διασύνδεση υπάρχει με αυτό. Διότι αν θεωρεί ότι ο κόσμο έχει δίκιο όταν συμφωνεί μαζί του, πείτε αντίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκέφτεστε έτσι. Πάει, ξεφανίστηκε. Και είμαστε στο δρόμο που δεν έχει επιστροφή. Αν θέλετε να σηκώνετε τα χέρια στον αέρα και να λέτε, ποφ, αν λέτε ότι ήταν επιτυχή αυτό που κάνετε μετά τον Brexit, μπορείτε το πείτε. Εγώ, η λύση μου είναι να σηκώνω τα χέρια στον αέρα. Δεν είναι απάντηση αυτή. Μιλάμε για το μέσο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν έχετε χρόνο, άλλο ένα λόγο είναι αυτό για τον οποίο ο κόσμο θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην παρετήσετε, μην σηκώνετε τα χέρια στον αέρα. Και ανοίξτε τα χαρτιά σα τα καταραμένα επιτέλου. Πείστε γιατί διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω αλαζονία αυτών που είναι εδώ σε αυτή την αίθουσα. Επίση, καταραίει και για άλλου λόγου που μπορεί να ε, επηρεάζουν αυτά που λέω. Οι άλλοι λόγοι θα αυτοθεραπευτούν. Εάν σταματήσετε να το παίζετε ανώτεροι και να έχετε τέτοια αλαζονία, θα διορθωθούν τα πράγματα. Ε, ναι, να πω κι εγώ ότι, ε, κύριε συνάδελφε, δεν έχουμε έρθει εδώ για να προσβάλλουμε τους ε, καλεσμένους μας. Αν κάποια πράγματα δεν μας αρέσουν, οι προσβολές δεν είναι λύση, διότι δεν οδηγούν πουθενά. Ο κύριος Στάς τώρα έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ιταλιάνερ, θα ήθελα να επανέλθω σε μια ερώτηση που από ό,τι θυμάμαι σας είχα θέσει και πέρσι. Όπως είπατε στην εισαγωγή σας, γνωρίζαμε ότι το 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού δαπανάται στη διαχείριση κοινής πολιτικής μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης η Επιτροπή Προπολογισμών εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα θυμάστε το Γιάνν Μουλντέρ, ήταν ένας από τους ανθρώπους ε, που ξεκίνησε την πρωτοβουλία μας πριν από κάποια χρόνια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λοιπόν ε, ε, ζητάμε να είναι υπόλογα τα κράτη-μέλη και να λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για τις δαπάνες. Και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποια δήλωση από τους Υπουργούς Οικονομικών της κάθε χώρας. δεν τα καταφέραμε ποτέ. τέσσερι χώρες και εν μέρη αποδέχτηκαν τις προτάσεις μας και τις υλοποίησαν. Οι περισσότερες από αυτές όμως είναι χώρες οι οποίες είναι αρκετά επιφυλακτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ενωμένο Βασίλειο, οι κάτω χώρες, η Δανία είναι χώρες λοιπόν οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο ε, ποσοστό ευρωσκεπτικισμού. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς λέτε ότι δεν λειτουργεί στο βέλτιστο δυνατό βαθμό η παρούσα πρακτική, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα και κάποια κράτη-μέλη απλώ οχυρώνονται πίσω από την ομοσπονδιακή του δομή. Ένα χρόνο μετά όμως, βλέποντας και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, διαπιστώνω ότι τα κράτη-μέλη θα έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζουν ότι κάποια ποσά ε, πληρώνονται χωρίς να υπάρχει λόγο. Κάποια, ε, κάποια κράτη-μέλη φαίνεται να το γνωρίζουν. Τι πρωτοβουλίες αναλάβατε εσείς στη διάρκεια του τρέχοντος έτους για να το διορθώσετε αυτό, για να διασφαλίσετε ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, ξοδεύονται ασυστόλως και ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και υπάρχει υπεύθυνη στάση ενώπιον της ε, ε, κοινοτική χρηματοδότησης. Δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως μάνα εξ η οποία φτάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να θεωρούν όλοι ότι λαμβάνουν δωρεάν αυτά τα χρήματα χωρίς να είναι υπόλογοι σε κανέναν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ιταλιάνο για τις πληροφορίες. Θα ήθελα και εγώ να ε, θέσω κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά την πολιτική και τη στρατηγική των προσφύγων που ε, γνωρίζω ότι έχετε και εξειδικευμένο προσωπικό στη Γενική σας Γραμματεία να ασχολείται με τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να μου πείτε τι εκτελεστική ικανότητα έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, τηρήσει τις συμφωνίες. Γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πλήρους απελπισίας. Από ό,τι λέει ο Επίτροπος υπάρχουν χρήματα, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά και αυτό το οποίο μας ε, ε, θέτουν οι πολίτες είναι ότι υπάρχει ε, πλήρης αδυναμία εφαρμογής και απορρόφησης αυτών των κονδυλίων. και μετά επιβάλλονται ε, τεράστια πρόστιμα ε, για, για κάποια πράγματα σήμαντα και γι' αυτό που είναι τόσο σημαντικό η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να ε, το εφαρμόσει όπως πρέπει. Επίσης, τι γίνεται με τους Ευρωπαίους ε, υπαλλήλους, τους Ε, έχουμε τις συνέπειες του Brexit, υπάρχει όλος αυτός ο λαϊκισμός και το θέμα της προβολής που έχουν οι ευρωσκεπτικιστές και οι ξενόφοβοι. Ε, τίθενται θέματα τύπου γραφειοκρατία ε, κλπ. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα λοιπόν που πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό. Τρίτον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία είναι η εξωτερική ανάθεση, το οποίο είναι πράγμα το οποίο πλήττει τις υπηρεσίες, γιατί επειδή δεν υπάρχουν δημόσιες θέσεις και πόροι, πρέπει να τα αναθέτουμε κάπου εξωτερικά αυτά. Και ε, από την άλλη, και όχι μόνο για θέματα ασφάλεια ε, και για λόγου αποτελεσματικότητα, υπάρχει μια τάση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εσωτεροποιούμε τι διάφορε υπηρεσίε. Εσεί λοιπόν πού στέκεστε όσον αφορά αυτέ τι δύο τάσει, οι οποίε είναι αρκετά αντιφατικέ μεν, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού στέκεται. Ε, επόμενο θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι πρέπει να ζητάμε περιοδικά από τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες και Οργανισμούς να μας λένε τι ακριβώς κάνουν σε αυτές τις δηλώσεις συμφερόντων. Πόσο ελέγχεται αυτό. Και τέλος, όσον αφορά την κινητικότητα των υψηλών αξιωματήχων, θα ήθελα να μας πείτε, για παράδειγμα, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ε, ε, Research, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής από το 2010, είναι Γενικός Διευθυντής σε μια κρίσιμη θέση, διότι είναι αρμόδιος για μια σειρά από πολύ σημαντικά προγράμματα πέραν του ορίζοντα 2020 και θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν εφαρμόστηκε η πολιτική κινητικότητα που εφαρμόζεται σε όλε τι υπόλοιπε γενικέ διευθύνσει. Απλώ για να γνωρίζω για ποιο λόγο γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο στη λίστα των ομιλητών, ο νέο μα συνάδελφο, κ. Σαφάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση που αφορά την γραμματεία της Όλαφ, του Οργανισμού Καταπολεμής των Απατών, διότι είναι προνόμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας να που κληρονομήθηκε πρόσφατα πριν η γραμματεία της Όλαφ εξασφαλιζόταν επί την Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ, αν θυμάμαι σωστά και αν άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν επειδή υπήρχε μεγάλη αφιβολία για τη δυνατότητα τη Επιτροπής Εποπτείας τη Όλαφ να σέβεται τον κανόνα περί ανεξαρτησίας που ισχύει για έναν οργανισμό κατά των απατών. Θα ήθελα να γνωρίζω πώς πηγαίνουν τα πράγματα όσον αφορά την αλλαγή. Θα ήθελα να ξέρω κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά το θέμα της ανεξαρτησίας που ισχύει για την Όλαφ. Θέτω το ερώτημα διότι πρόσφατα ε, μια έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας όσον αφορά τις ανεξάρτητες, τους ανεξάρτητους διοικητικούς φορείς που αφορούσε τις αρχές της διοικητικές της ανεξάρτητες στη Γαλλία είχε ένα κείμενο για την, μια αναφορά στην Όλαφ αρνούμενη την ιδιότητα της διοικητικής ανεξαρτησίας βάσει των κριτηρίων της γαλλικής κυβέρνησης και της γαλλικής διοίκησης. Ο κ. Φλάνναγκαν για άλλη μια ακόμα φορά. Κυρία Πρόεδρε, μιλήσατε για προσβολή κατά ανθρώπων. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Το πιο προσβλητικό που άκουσα εγώ στη ζωή μου ήταν η ιδέα ότι 70 εκατομμύρια άνθρωποι, ε, τους λένε 70 εκατομμύρια ανθρώπους, κάνατε λάθος. Ήταν μια απόφαση που πήραν αυτοί οι άνθρωποι να προχωρήσουν. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπατε είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα θα αντιμετωπίσει το Brexit. Δεν θα γίνει τακτικό το Brexit, δεν θα επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα εξασφαλιστεί ότι θα σπρώξουν κάτω στο λαιμό των Βρετανών ότι έκανα λάθο. Έτσι πιστεύω. Και αν κάποιος προσβάλλεται από αυτά που λέω, τότε αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει κάτι για αυτό, για τη σύγκρουση των συμφερόντων. Πρέπει να κάνει κάτι για το ότι δεν δέχεται τη βούληση των λαών. Εάν δεν το κάνει αυτό, χάθηκε. Και αν προσβάλλεστε από αυτό που λέω, τι να σας πω, να πάψετε να προσβάλλεστε, αντιμετωπίστε το πρόβλημα. Και τότε θα λυθούν τα προβλήματα, να σταματήσετε να προσβάλλεστε. Όχι, όχι, συνάδελφε, μην μπλέκουμε τα αίτια με τα αιτιατά. Υπάρχει το κατάλληλο βήμα για τις ε, κατάλληλες τοποθετήσεις. Εγώ δεν αναφέρθηκα στο περιεχόμενο, αναφέρθηκα στον τρόπο σας. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Έχω μπει και ίδια στον κατάλογο των μιλητών. Όχι, όχι κύριε συνάδελφε, δεν θα κάνουμε τώρα εδώ συζήτηση. Αν μας μένει χρόνο στο τέλος, αλλά δεν το βλέπω. Ε, Τέλο πάντων, να πω παρεπτόντω ότι ο κύριο Γενικό Γραμματέα ήταν εδώ στι 9. Εμεί δεν ήμασταν εδώ στι 9. Γι' αυτό λοιπόν α δείξουμε λίγη κατανόηση, α κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα και α δώσουμε στου ε, καλεσμένου μα την ευκαιρία να απαντήσουν. Εγώ έχω κάποιε ερωτήσει λοιπόν. Εξή, μόχλευση των δημοσιονομικών ε, μέσων. Μα είπατε για το 2,9% ε, το οποίο θα τλήθει από ξένα κεφάλαια. Ε, τι ακριβώ εννοείται με ξένα κεφάλαια αν χρησιμοποιήσουμε μόνο δημόσια κονδύλια, τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ε, ο σαφής ορισμός της μόχλευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο χρήμα. Ε, αυτό ίσως χρειαστεί να το συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα νούμερα που έχετε υπόψη για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Έπειτα, κώδικας δεοντολογίας πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι επίτροποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν βλέψεις για άλλο ανώτερο πόστο και δεν θα γίνουν, για παράδειγμα, λομπίστε σε δύο-τρία χρόνια ή δεν θα του χρησιμοποιήσουν. Αυτό με ανησυχεί, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος μηχανισμός που να φροντίζει να κάνει αυτού τους ελέγχους. Και ναι, πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κατάχρηση, να χρησιμοποιήσουν τέλο πάντων ορισμένοι την θέση τους έτσι ώστε να βελτιώσουν τη μελλοντική τους ε, κατάσταση. Το είδαμε στην προηγούμενη Επιτροπή. Μετά να πω ότι με ανησυχεί κάπως ε, το ότι πουλάμε την ε, αλλαγή του Omnibus ως ε, μεγάλο πίτευμα, απλοποίηση κτλ. Εγώ πιστεύω πως τα πράγματα περιπλέκονται ακριβώς για να μην αλλάξουν και νομίζω πως η διαδικασία που ακολουθείτε δεν είναι δίκαιη. Βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση χρόνου. Ε, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές χωρίς εκτίμηση αντικτύπου. Πού είναι η εκτίμηση αντικτύπου για αυτές τις ε, προτάσεις οι οποίες είναι λεπτομερέστατες, πάνε πολύ μακριά ε, για τα δημοσιονομικά μέσα. Ε, εσείς μας λέτε πως ε, γίνονται πιο απλά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Πιστεύω πως αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει ο κόσμος γύρω μας. Ε, και θα αλλάξουν οι συνθήκες και για τους επενδυτέ και για τους καταθέτε. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, απλουστεύουν τα πράγματα για ποιον όμως δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μας πουληθεί με πολύ ωραία λόγια κάτι το οποίο θα κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη. Ε, και για τις διαβουλεύσεις σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας να πω πως αυτή τη στιγμή προσπαθούμε, δεν έχουμε όμως καταφέρει να πείσουμε όλους ε, τους ε, συναδέλφους για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας αλλαγής. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτό, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα. Ε, τώρα θα σας δώσω πάλι το λόγο για τις απαντήσεις. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής για τις ερωτήσεις που έθεσαν και τα θέματα που έθεξαν. Επί Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Ε, κάποιες ε, ερωτήσεις ήταν ε, εγγενώς πολιτικές, δεν είναι στις αρμοδιότητές μου αυτό, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Ετέθη μια γενική ερώτηση όσον αφορά τον ιδιωτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παρούσα χρονική συγκυρία. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ ευθύς εξ αρχής, μόλις ανέλαβε καθήκοντα, προσπάθησε να ασκήσει ηγετικό ρόλο αναγνωρίζοντας ότι ε, αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ασχολείται με την κάθε ανθιπολεπτομέρεια της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρότεινε τις 10 προτεραιότητές του, οι οποίες είναι ε, πολύ συγκεκριμένε. Αν δείτε τις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις νομοθετικές προτάσεις, ε, ε, έχουν μειωθεί οι προτάσεις κατά 40% κατά μέσο όρο. Ε, υπήρχε και μία ε, ερώτηση για τη σχέση ε, με το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν νομίζω ότι είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν θα σεβαστεί τη βούληση των Βρετανών πολιτών. Είπαμε απλώς ότι η αποχώρηση που επιθυμεί ο Βρετανικός λαός θα πρέπει να γίνει με όσο το δυνατόν πιο ομαλό τρόπο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. έγιναν αρκετές ερωτήσεις ε, για τον κώδικα διοντολογίας. Να πω ότι υπάρχουν δύο θέματα όσον αφορά τον κώδικα διοντολογίας. Πρώτον είναι κώδικας και δεύτερον αφορά την διοντολογία. Η διοντολογία εξορισμού είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ε, περιοριστεί σε κανόνες. Υπάρχει όμως και το άρθρο 245 της συνθήκης. Ε, αναπόφευκτα λοιπόν θα υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση κατά πόσον μια συμπεριφορά είναι σωστή ή όχι. Και νομίζω ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ ήταν απόλυτα σαφής ως προς την άποψή του για τις νέες δραστηριότητες ε, του προκατόχου του. Το κατά πόσον ε, αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται νομικώς είναι άλλο θέμα συζήτησης. Δεν μπορούν να προβλεφθούν τα πάντα από τους κανόνες. Αλλά υπάρχει μια σαφέστατη σύσταση από τις διεθνείς οργανώσεις ότι εάν είναι μεγαλύτερη η διάρκεια αυτής της περίοδου cooling off ε, μεταξύ δύο διαφορετικών ε, ε, θέσεων θα μειωθεί ο αριθμός ε, των ανθρώπων που κατήχαν προηγουμένως δημόσια αξιώματα ε, και τώρα εργάζονται για άλλα συμφέροντα. Και επομένως γι' αυτό έχει προτείνει και ο, ο πρόεδρος Γιούνκερ αύξηση αυτών των περιόδων αργίας, αν θέλετε, από τα τρία στα τέσσερα χρόνια. εξεπλάγει από τα σχόλια που έγιναν για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το άγχος που διακατέχει τον εργασιακό τους βίο. Κάποιος είπε ότι το προσωπικό ε, έχει όλο ένα και περισσότερε ε, θέσει εργασία. Ναι, η Γενική Γραμματεία έχει περισσότερε θέσει εργασία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά ε, για πέντε χρόνια, για μία πενταετία, είχε μία μείωση τη τάξη του 1%, η οποία εφαρμόστηκε και παρόλα αυτά οι προκλήσει ε, δεν σταμάτησαν να αυξάνονται. Εσωτερικώ λοιπόν ανελήφθησαν μία σειρά από πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίε όσον αφορά την εφημερία. Ε, του προσωπικού, ενθαρρύνουμε το προσωπικό να είναι σε καλή φυσική κατάσταση στο χώρο της εργασίας και σε μια πρόσφατη έρευνα προσωπικού που έγινε, οι απαντήσεις όσον αφορά την ευημερία του προσωπικού ήταν θετικές. Σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον υπάρχουν λοιπόν κάποια ενθαρρυντικά ε, στοιχεία. Ε, δεν ε, σας κρύβω βέβαια ότι είναι ε, αγχώδης η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, κυρίως όσον αφορά την ισορροπία εργασιακού βίου και οικογενειακού βίου, χρησιμοποιούνται μέθοδοι τηλεεργασίας κλπ. Σε μια ερώτηση τώρα για την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπηρεσιών και την ερώτηση που έκανε ο εισηγητής του προηγούμενου έτους. Θεωρώ προσωπική μου ευθύνη πέραν όλων των ομάδων ε, προγραμμάτων ε, των οποίων προεδρεύουν τώρα οι αντιπρόεδροι γιατί οι αντιπρόεδροι προεδρεύουν σε όλες αυτές τις project teams ε, κάνουμε ακριβώς το ίδιο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Δεν έχει αναλυφθεί καμία πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία να μην υπόκειται σε έντονη συνεργασία προς τα πάνω στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν από 10 χρόνια δεν εργαζόμασταν με αυτόν τον τρόπο. Πολλές πρωτοβουλίες ε, ε, ε, προετοιμάζονταν μεμονωμένα και από εκεί και πέρα το γεγονός ότι οι υπηρεσίες τώρα υποχρεούνται να έχουν μια διοργανική ομάδα κατά την προετοιμασία της νέας πρότασης και πολύ συχνά προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Παρεπιπτόντων. Δεν προεδρεύουν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις, αυτό αποτέλεσε μεγάλη αλλαγή για τη συνεργασία εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια είχαμε μια ερώτηση για την ε, πρόσβαση σε, φον, σε πόρους του ε, σχεδίου Juncker. Όπως σας είπα, η γενικότερη απορρόφηση του σχεδίου Juncker είναι πάρα πολύ καλή και έχουμε προσελκύσει και πολλές ιδιωτικές επενδύσεις από το συνολικό πεσό το οποίο διδασμεύτηκε το Δεκέμβριο πέρσι περίπου το 90% ε, χρηματοδότησε ε, εκτός ε, προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπήρχε και πολύ μεγάλη μόχλευση εντός του Ταμείου Juncker. Και πώς μπορεί να γίνει αυτή η μόχλευση διότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό επιτρέπουν ε, να προσφέρουμε εγγυήσει στους επενδυτές. Επομένω, υπάρχει κάλυψη για το πρώτο τμήμα της απώλειας που μπορεί να περιλαμβάνει μια επένδυση και αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο για τους ε, ιδιώτες επενδυτές ε, προκειμένου να επενδύσουν στα σχέδια αυτά. Μετά. Ετέθη μια ερώτηση για την επικουρικότητα, τους γενικότερους κανόνες επικουρικότητας. Στις αξιολογήσεις αντικτύπου που κάνουμε, συνήθως αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που τίθεται. Κατά πόσον η αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία τώρα έχει αντικατασταθεί και από το ε, Συμβούλιο ρυθμιστικού ελέγχου θα δείτε ότι υπήρχαν και κάποιες ε, περιπτώσεις στις οποίες απορρίφθηκαν οι ε, αξιολογήσεις επιπτώσεων και είναι αρκετά υψηλός αυτός ο αριθμός. Και είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Εν και μια ερώτηση για την ε, κρίση των προσφύγων και την ε, εκτελεστική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό το επίπεδο. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι η προσφυγική κρίση αποτελεί συγκεκριμένο παράδειγμα του τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να, πώς πρέπει να συνεργαστεί επιτόπου με τα κράτη-μέλη. Σε αυτή την περίπτωση με την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ο Γενικός Διευθυντής που είναι υπεύθυνο ε, για την υπηρεσία υποστήριξης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μεταβαίνει στην Ελλάδα δύο ημέρες την εβδομάδα περίπου για να βοηθήσει τους Έλληνες ε, υπαλλήλους επιτόπου για την αντιμετώπιση της χρήσης, ε, προσφέρει συμβουλές για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό παράδειγμα του πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και όχι απλώς να εκδίδουμε ένα σύνολο κανόνων, αλλά να υπάρχει ε, πραγματική συνεργασία επιτόπου. Βεβαίως ε, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής που τώρα έχει 1500 άτομα προσωπικό, επιχειρησιακό προσωπικό ε, είναι και αρμόδια για την βοήθεια προς τα κράτη-μέλη για την εξασφάλιση των εξωτερικών συνόρων η κυρία Γιάλα Σέντερ ρώτησε και για την εξωτερική ανάθεση αλλά και την εσωτερική ε, αντιμετώπιση των διαφόρων υπηρεσιών. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι εξωτερική ανάθεση. Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται τα τελευταία δέκα χρόνια είναι η σύσταση εκτελεστικών υπηρεσιών. Ε, θεωρώ ότι λειτουργεί πολύ αποτελεσματικό αυτό και αυτές οι υπηρεσίες συνεργάζονται πάρα πολύ καλά με τις ε, αδελφές γενικές διευθύνσεις. Όσον αφορά την κινητικότητα των ε, ανώτατων αξιωματούχων, ε, έχουμε συγκεκριμένους ενδεικτικούς κανόνες για τα θέματα κινητικότητας, αλλά αν υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν ε, ε, ένα σημαντικό πόστο το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν υπάρχει υποχρέωση κινητικότητάς τους ε, μόνο για λόγου κινητικότητας. Ο προκάτοχός μου, για παράδειγμα, είχε την ίδια θέση για 10 χρόνια. Ελπίζω εγώ να μην παραμείνω εκεί τόσο πολλά χρόνια, αλλά είναι γιατί είναι αρκετά δύσκολη δουλειά, αλλά αυτό είναι τελείως προσωπικό σχόλιο. Ε, κατόπιν ετέθη μια ερώτηση για τη γραμματεία της ε, Εποπτικής Επιτροπής της Όλαφ. Όπως έχει ανακοινώσει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θα μεταφερθεί αυτή η υπηρεσία εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα βρίσκεται σε μια ουδέτερη υπηρεσία ώστε να διασφαλίζεται και η ανεξαρτησία της λειτουργίας αυτής της Εποπτικής Επιτροπής. Ε, υπήρξε και μια ερώτηση για την ανεξαρτησία της ίδιας της Όλεφ, αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση. Νομίζω ότι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες της Όλαφ γίνονται εντελώ ανεξάρτητα. Και τουλάχιστον από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν αμφισβητεί κανείς ε, την ανεξαρτησία της Όλαφ. Κυρία Πρόεδρε, προσπάθησα να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Α, συγγνώμη, την ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έχετε δίκιο. Θα ζητήσω από τον συνάδελφο, τον κύριο Κάφ, να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για τη λογοδοσία των κρατών μελών όσον αφορά την κοινή διαχείριση οι εθνικές δηλώσεις που υπεγράφησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Σουηδία και τη Δανία, αυτό πήρατε σαν παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου και των κρατών μελών καθόρισαν κριτήρια για το πώς να χρησιμοποιήσουμε τις διαβεβαιώσεις που παρέχονται σε εθνικές δηλώσεις. Ε, Δυστυχώ, η επιτυχία δεν ήταν πολύ μεγάλη, όπω γνωρίζετε. Αντί τέσσερις έχουμε τρία κράτη-μέλη που υποβάλλουν εθνικές δηλώσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο σταμάτησε από ό,τι γνωρίζω, όμως συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να αποφύγουμε τα σφάλματα, χρησιμοποιούμε εργαλεία, όχι μόνο σεμινάρια και κατάρτιση, αλλά διακοπές και αναστολές πληρωμών, όποτε υπάρχει ένα εντοπιστέν σφάλμα ή σύστημα που εντοπίζεται έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε οικονομικές διορθώσεις και το κάνουμε αυτό τακτικά. Και οι πληροφορίες παρέχονται στην ανακοίνωση για την τη σχετική κοινοποίηση, ανακοίνωση μάλλον για την προστασία των οικονομικών συμφωνών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δύο συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και τους παρακαλώ να είναι πάρα πάρα πολύ σύντομοι. Ε, πρώτος το λόγο έχει ο κ. Μάιρς. Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω τον ε, κύριο Γενικό Διευθυντή. Αναφέρθηκε στα θέματα της ε, συνοριοφυλακής, ε, ιδίως σε σχέση με την Ελλάδα. Και θα ήθελα να το ρωτήσω γενικότερα, ε, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία τεράστιας καθυστέρησης στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου, οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα. Ήθελα να μου πείτε με στοιχεία όταν ξεκίνησε η διαδικασία της ε, κοινή δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας είχε υποσχεθεί ο κύριος Γιούνκερ ότι θα πάνε τουλάχιστον 400 εμπειρογνώμονες σε θέματα παροχής ασύλου. Επίσης 400 νομικοί. Μέχρι στιγμής έχουν πάει ελάχιστοι και αυτό που γίνεται είναι να έχουμε μια υπερσυγκέντρωση προσφύγων και παρανόμων μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου και να υπάρχει ασφικτική κατάσταση. Έχετε κάποια στοιχεία για το πώς έχει εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Δεύτερη σύντομη παρατήρηση. Αναφερθήκατε για τη συνεργασία της Κομισιόν με τις ελληνικές αρχές. Αυτή η συνεργασία γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο πλαίσιο του μνημονίου, δηλαδή η συνεργασία της Κομισιόν ως Τρόικα με την ελληνική κυβέρνηση. Και μια παρατήρηση προς τη Γραμματεία ε, επειδή, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει διερμηνία στα ελληνικά, το βλέπω, όμως ε, δεν υπάρχει η μετάδοση της συζήτησής μας μέσω το Web TV του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ελληνικά. Αν βάλετε δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Επομένως θα ήθελα να το ρυθμίσετε αυτό, διότι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση την παρακολουθούν στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες. Αν μπορεί να ρυθμιστεί, γιατί το ήλεγξα και δεν μπορεί να κάνει κανείς επιλογή από μακριά να ακούσει τη συνεδρίαση στα ελληνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρατήρηση αυτή ε, και για τα σχόλιά σας. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρατε, ότι, τον Μισελ Μπαρνιέ και ότι ε, θα ήθελε το Brexit να λάβει χώρα με τρόπο ήπιο και ε, φυσιολογικό. Στο Στρασβούργο είχα την δυνατότητα να συναντηθώ με τον Μισελ Μπαρνιέ και αυτό που κατάλαβα από τη συνάντησή μας είναι ότι δεν κατάλαβε αυτά που λέγαμε, ε, γιατί τα αγγλικά του δεν ήταν επαρκή. Εσείς βλέπω πως ε, έχετε άπτεστη γνώση των αγγλικών και, το, και ο συνεργάτης σας επίσης. Βασικά βλέπω πως τα αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω, ε, δεδομένου ότι θέλετε το Brexit να γίνει ομαλά, θεωρείτε πως μια αγγλόφωνη χώρα θα μπορεί να διαπραγματευτεί ε, ενδεχομένως με βοήθεια διερμηνέα, με κίνδυνο να χαθούν λεπτομέρειες. Γιατί να μην επιλέξουμε έναν αγγλόφωνο, ένα φυσικό ομιλητή της εγγλικής ε, για διαπραγματευτή ο προκάτοχός, ε, ή προκατοχός σας μάλλον είπε σε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο της Ιρλανδίας ότι γιατί να μην αρχίσουμε να μιλάμε γαλλικά ας πούμε γερμανικά, να ξεφύγουμε από τη Μεγάλη Βρετανία. Εγώ πιστεύω πως κάναμε ένα λάθος, πως ε, αποχωρήσαμε από την πρώτη συνάντηση συγχυσμένοι, μπερδεμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Σταλιάνερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομο θα είμαι σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για τα αιτήματα ασύλου. Να πω πως αυτό απαιτούσε την δημιουργία των κατάλληλων δομών και διαδικασιών από την ελληνική πλευρά. Μαζί με τη στήριξη εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη. Υπήρξαν καθυστερήσει και από τις δύο πλευρές και συνεχίζουμε να κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη για να στείλουν προσωπικό, να στείλουν εμπειρογνώμονε για να στηρίξουν τις ελληνικές αρχές. Ε, μπορώ να σας δώσω στοιχεία, αλλά αν προτιμάτε θα το κάνω διμερός ε, και τότε θα σας δώσω τα συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα για το πλαίσιο της ε, Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και την Τρόικα η στήριξη που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πηγαίνει προς τις, ε, την υπηρεσία ε, στήριξης διαθερωτικών μεταρρυθμίσεων. Είναι ένα κομμάτι του γενικότερου πλαισίου συνεργασίας με τα κράτη-μέλη, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με όποιο άλλο κράτος μέλο ζητήσει βοήθεια. Και νομίζω πως όπως είδαμε σε αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε οποιαδήποτε γλώσσα χρειάζεται εξαιτία της εξαιρετικής δουλειάς των διερμηνέων. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα στον εισηγητή το λόγο για να κλείσουμε. Είπαμε ήδη πως δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Η συζήτηση ήταν περιεκτικότατη. Να ευχαριστήσω ξανά τον κύριο Ιταλιάνερ για την παρουσίασή του και τους συναδέλφους όλους για τις τοποθετήσεις τους. όλη η συζήτηση νομίζω πως θα αντικατοπτριστεί στην έκθεση για την απαλλαγή. Κύριε Ιταλιάνερ, αναφέρατε πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν και εμάς, το ΕΦΣΙ για παράδειγμα, τα δημοσιονομικά μέσα, το ε, καταπίστευμα, πώς θα λειτουργήσει. Όμως θεωρώ πως ε, μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις θα καταβάλουμε τις κατάλληλες προσπάθειες για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας ξαναδούμε κύριε Ιταλιένερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας και για τις γραπτές απαντήσεις. Και θα ήθελα τώρα ε, να παρακαλέσω όσους δεν είναι μέλη της Επιτροπής ή όσους δεν έχουν θέση εδώ να αποχωρήσουν διότι θα, θα συνεχίσουμε με το κοινό σημείο με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Για την επόμενη ώρα το σημείο αυτό θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ να καταλήψετε την αίθουσα όσοι δεν...